Κυρίες και κύριοι, αποτείουμε φόρο και θυμόμαστε απόψε τους ανθρώπους εκείνους που πριν από 20 χρόνια στις φαγές στην πόλη Σρέμπνενιτσα δολοφονήθηκαν. 8.000 νέοι και